Είμαι και πρόθυμοι να αναλάβουμε οποιαδήποτε βήματα και διαβήματα σε σχέση με τι αρχέ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για να επιληθεί το πρόβλημα. Αυτό ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ, Επίτροπε. Έχουμε 7 προτάσει ψηφίσματο που θα ψηφιστούν σήμερα στην Ολομέλεια στι 11.30. Περνάμε στο επόμενο σημείο, στην ημερήσια διάταξη. Η περίπτωση των κοριτσιών στο Πακιστάν. Ιδιαίτερα η περίπτωση τη ε, Μαλάλα Ιουσαφσάη. Για 1,5 λεπτό θα λάβει τον λόγο η κυρία Κάβης. Η Μαλάλα Γιούσφα επλήγει από τους ε, Ταλιμπάν. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η κατάσταση των γυναικών στο Πανιστάν. Είναι η τρίτη πιο επικίνδυνη χώρα στον ε, κόσμο. Είναι Ισλαμική χώρα, αλλά στην ουσία αντι-Ισλαμική. Οι Ταλιμπάν ε, πλήττουν τις, και τιμωρούν τις γυναίκες στο Πακιστάν και στο γειτονικό Αφγανιστάν. Δεν τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να ε, ζήσουν τη ζωή τους. Η τραγωδία της ε, Μαλάλα κλειδώνησε και κλώνησε τον κόσμο, ακόμα και το ίδιο το Πακιστάν. Το μόνο έγκλημα αυτού του κοριτσιού ήταν να απαιτήσει τα δικαιώματά της, δικαίωμα στην εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να λέμε business as usual με το Πακιστάν. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Θα πρέπει οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές να απαλλαχθούν από αυτό το είδημα που λέγεται Ταλιμπάν και να καταπολεμήσουν την μισαλοδοξία που πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προβαίνει σε συμφωνίες συνεργασίες με μια κυβέρνηση η οποία αρνείται τα πάντα. Τη στιγμή που χτυπά παιδιά επειδή πηγαίνουν στο σχολείο, που χρησιμοποιούνται τα παιδιά ως ε, μορφή αντιπραγματισμού ή δημιουργούν ή χρησιμοποιούνται από τους Ταλιμπάν σε επιθέσεις αυτοκτονίας. Η κοινωνία των πολιτών είναι ανύπαρκτη. Γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Προβέρα ε, ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε απαράδεκτη, απαράδεκτη κατάσταση, εσχημοσύνη, ασχημοσύνη, εδώς, αυτό θα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίζει την περίπτωση της ε, ε, Μαλάλα. Η Μαλάλα ήθελε απλώς να πάει στο σχολείο, τίποτα άλλο. Γι' αυτό την ε, πυροβόλησαν στο κεφάλι και στην πλάτη. Αυτό το εγχείρημα των Ταλιμπάν στην ουσία τι κάνει. Θέλει να διαγράψει ανθρώπινα δικαιώματα ουσίας. Η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτό μας λέει. Αυτό είναι το πρότυπο ζωής που προτείνουν οι Ταλιμπάν στο μουσουλμανικό κόσμο. Ε, μη σεβόμενη τη ζωή των άλλων. Βεβαίως καταδικάζουμε αυτές τις δειλές ε, και σκληρές πράξεις, θα θέλαμε όμως όλο, ολόκληρο το Ισλάμ να καταδικάσει αυτά τα εγκλήματα. Δεν μπορούμε να σιωπούμε. Αυτό σημαίνει ότι συμμεριζόμαστε και είμαστε συνένοχοι και αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστούμε κύριε Προβέρα. Η κυρία ναι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα συζητάμε το θέμα της Μαλάλα Γιουσουσάη. Μία 14χρονη από την κοιλάδα Σουέτ στο Πακιστάν, η οποία στις 9 Οκτωβρίου πυροβολήθηκε στο λαιμό και στο κεφάλι πηγαίνοντα στο σχολείο. Τραυματίστηκε σοβαρά. βεβαίω και θα την στηρίξουμε και θα συμπεριφερθούμε συμπαρασταθούμε στην ίδια και στην οικογένειά της. Αυτό φαίνεται και από το ψήφισμα. Οι Ταλιμπάν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση και ε, ξέδωσαν και μία δήλωση πως θα προσπαθήσουν να την ξανασκοτώσουν αν ανακάμψει από τα τραύματά της. Ξέρετε τι περνάνε τα κορίτσια στη χώρα αυτή. Βία στο σπίτι, δεν πάνε σχολείο, ε, υποχρεώνονται να παντρευτούν. Η βία κατά των κοριτσιών στα, στο Πακιστάν δεν διώκεται. Πιστεύω πως όταν τα παιδιά γίνονται στόχος ε, τέτοιων στρατιωτικών επιχειρήσεων και αυτό γίνεται αποδεκτό από την κυβέρνηση της χώρας, το καθεστώς δεν έχει μέλλον, τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδεύονται καλύτερα από τους γονείς τους και εάν οι θείοι τους και οι πατεράδες τους και οι αδελφοί τους δεν τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν το βασικό δικαίωμα στην παιδεία, αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Ένα λεπτό παρακαλώ, ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι μόνο ένα προηγούμενο αυτό. Δεν είναι μια εξαίρεση αυτό το προηγούμενο παρότι είναι ιδιαίτερα οδυνηρή, επώδυνη περίπτωση είναι μια περίπτωση που κατά κανόνα επαναλαμβάνεται διαρκώς και αδιαλείπτως όχι μόνο σε αυτή τη χώρα αλλά σε όλη την ευρύτερη περιφέρεια ένα πράγμα θα έπρεπε να είναι σαφές για όλους ότι θα έπρεπε διαζώσεις ε, και κάθετα να πούμε τι συμβαίνει εδώ. Ένα μέρος αυτής, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας αυτής αποδέχεται, δέχεται τους Ταλιμπάν και τις πράξεις και τις τακτικές τους. Αυτό είναι το δράμα, η δραματική κατάσταση στο Πακιστάν, διότι αυτό θα έχει επιπτώσεις για το μέλλον αυτής της χώρας και το μέλλον των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Θα ήθελα λοιπόν και έναντι των εταίρων μας, όχι μόνο στην Ευρώπη, να καταστήσουμε σαφές ότι εκείνοι που διαπραγματεύονται με τους Ταλιμπάν, ιδιαίτερα εκείνοι που διαπραγματεύονται με τους Ταλιμπάν, να γνωρίζουν το τι συμβαίνει διότι πολλές φορές εξυπηρετούν τα πολιτικά του συμφέροντα και όχι τα δικαιώματα του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ. Κυρία Λάμπερτ, παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τον Πρόεδρε. Είδαμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να αντισταθεί κανείς κατά τον Ταλιμπάν όταν ο ίδιος προσωπικά η οικογένειά σου, οι δικοί σου οικοί και συγγενείς απειλούνται και δολοφονούνται κιόλα. μπορούμε στο Κοινοβούλιο πραγματικά να επενέσουμε την γενναιότητα της Μαλάλα και άλλων. Αυτά τα κορίτσια και αυτά τα αγόρια που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα σε αυτά τα σχολεία ακόμα και όταν απειλούνται από τους Ταλιμπάν υπήρξε μια πολιτική και δημόσια κατακραυγή στο ίδιο το Πακιστάν για αυτά τα τραγικά συμβάντα και θα έπρεπε να υποστηρίξουμε τις κραυγές αυτών των ανθρώπων που διαμαρτύρονται υπήρξαν αλλαγές στην νομοθεσία του Πακιστάν. Τώρα το πρόβλημα θα είναι η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, η υλοποίηση όλων αυτών. Διότι πολλοί θεωρούν, οι Ταλιμπάν θεωρούν ότι αυτή η μόρφωση, η παιδεία των γυναικών είναι απειλή για τις ίδιες τις δομές εξουσίας τους. Είδαμε επιθέσεις στην ίδια αυτή την περιοχή του Πακιστάν εις βάρος ε, των μαθητών, των κοριτσιών. Είναι κέρια σημασία να επενδύσει η κυβέρνηση στην δημόσια εκπαίδευση και παιδεία υπέρ αυτών των παιδιών να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ορθώσουμε το ανάστημά μας κατά των δυνάμεων της καταστολής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια ο κύριος ε, Μπένιαμιν, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το κατεπήγον ψήφισμα από διαφορετικές πολιτικές ομάδες ε, στοχεύει να καταδικάσει αυτά τα οποία έγιναν από τους ε, Ταλιμπάν. Πρώτον θέλω να δραχτώ της ευκαιρίας να συγχαρώ για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και περίθαλψης επιτόπου για το κορίτσι αυτό την Μαλάλα και που ε, πήγε στην Βρετανία. Η εκστρατεία για το δικαίωμα των κοριτσιών των, ε, να μπορούν να εκπαιδεύονται συγκίνησε ε, παγκόσμια και κάποιοι ακολουθούν την πρακτική των παιδικών γάμων. Οι γονείς φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους ιδιαίτερα τα κορίτσια στο σχολείο. Απευθύνται έκκληση ώστε η κυβέρνηση του Πακιστάν να παράσχει το δικαίωμα της ε, πρωτοβάθμιας εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν και τα θέματα των μεντρεσέδων, δηλαδή των ε, ιεροσπουδαστηρίων ε, και πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών στην εκπαίδευση. Δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει στο, στο Πακιστάν και την κυρίαρχη κυβέρνησή του το τι θα πρέπει να κάνει. Αλλά πώς μπορεί να πιστεύει κανείς ότι δικαιούται να σκοτώσει ένα κορίτσι επειδή πηγαίνει σχολείο. Μόνο οι αν υιοθετούν αυτή την άποψη και αυτό είναι καταδικαστέο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριος Μέρφυ παρακάτω. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω ε, την, το θαυμασμό μου για τη γενναία της ε, απόφαση να πάει σχολείο. Αυτή η επίθεση των Ταλιμπάν δείχνει πόσο δύσκολη είναι η ζωή των νεαρών κοριτσιών στο Πακιστάν. Είναι το τρίτο πιο επικίνδυνο κράτος για τις γυναίκες στον κόσμο. Κατοντάδες σχολεία έχουν καταστραφεί από ε, ακραίες, ακροδεξιές Ισλαμικές ομάδες που αυτή τη στιγμή ισχυροποιούν τη θέση τους στην κοινωνία. Και αυτό είναι τραγικό για τις γυναίκες ε, που φέρουν το βάρος της κατάρρευσης της συνεχιζόμενης της πακιστανικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε ε, τα όσα συμβαίνουν στο Πακιστάν να τα χωρίσουμε από τα όσα συμβαίνουν στην Αφγανιστάν. Έχουμε τις ε, οπισθοδρομικές ομάδες των Ταλιμπάν που δεν πρέπει να μην συνδεθούν με την ε, κατοχή του Αφγανιστάν από τους Αμερικανούς και τα πολεμικά γεγονότα που έχουν στοιχήσει τη ζωή σε 3.000 άτομα. Αυτή ε, από τα θύματα το ποσοστό των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους από τους 3.000 που ανέφερε είναι μόνο το 2%. Αντίθετα οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν ενισχύσει την ε, προσάρτηση ατόμων σε κάποιες ομάδες. Άρα λοιπόν η κατοχή του Αφγανιστάν θα πρέπει να λήξει. Περνάμε τώρα στις ομάδες. Έχουμε με μπλε κάρτα. Κύριε Μέρφυ, δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Τάνοκ. Κύριε Τάνοκ. Κύριε Μέρφυ, μπορείτε να με εξηγήσετε λοιπόν ποια είναι αυτή η κατοχή του Αφγανιστάν από την ΣΥΠΑ ε, έτσι όπως τη χαρακτηρίζετε εσείς ε, που εν είχε ως σκοπό να ε, απαντήσει στο θάνατο 3.000 ατόμων στους δίδυμους πύρους σχετίζεται με μια επίθεση κατά ένας νέο κοριτσιού γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν σχετίζονται εξηγήστε το μας παρακαλώ Μπορώ να το εξηγήσω αρκετά εύκολα. Έχουμε λοιπόν αυτή την έκθεση από την νομική η, αυτή η σχολή στη ΣΥΠΑ που λέει πως η ένταξη νέων μελών σε αυτές τις νέες τις ομάδες έχουν να κάνουν με τις επιθέσεις των Αμερικανών όπου ε, στην πραγματικότητα οι δυνάμεις αυτές των Ταλιμπάν επίσης επιτίθενται σε σχολεία και προσπάθησαν να σκοτώσουν τη Μαλάλα. Αυτή την πραγματικότητα αναγνωρίζω και Πιστεύετε πως η επίθεση και η συνεχιζόμενη κατοχή του Αφγανιστάν σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την επίθεση της 11 η Σεπτεμβρίου γιατί έχει φανεί ξεκάθαρα πως ε, δεν υπάρχει σύνδεση και μάλιστα υπήρχε ήδη ε, σχέδιο πριν την επίθεση για να γίνει αυτό στο Αφγανιστάν. Η κυρία Κορόλα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Με την εργασία που παρακολουθήσαμε, το έργο που παρακολουθήσαμε και σε σχέση με την Μπέναζιρ Μπούτο υπέρ του εκδημοκρατισμού του Πακιστάν που είχε επισκεφθεί το Ευρωκοινοβούλιο πρωτού ε, ε, δολοφονηθεί. Γνώριζε ότι θα την δολοφονούσαν, όμως ε, κατέβαλε κάθε προσπάθεια και σε αυτή την περίπτωση με αυτό το κορίτσι την ε, Μάλαλα βλέπουμε πόσο, ε, πώς εκφράζεται η αλληλεγγύη και στο Πακιστάν και αλλού. Βλέπουμε εδώ ότι ε, αποτέλεσε στόχο αυτό το κορίτσι. Πρόκειται για το δικαίωμα στην παιδεία και στην εκπαίδευση και είναι σημαντική υπόθεση αυτή, αυτό σε μια χώρα που έγινε η προσπάθεια από πλευράς ε, της ε, Μαλάλα να ε, εκπαιδευτεί. Έκρυβε τα βιβλία της, κρυφά διάβαζε επειδή είχε απαγορευτεί από τους Ταλιμπάν αυτό. Πολλά παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια δεν μπορούν να πάνε σε σχολεία και αυτό λόγω της πολιτικής και των απειλών των Ταλιμπάν. Και το Πακιστάν έχει μια νέα ηρωίνα που πραγματικά απέδειξε με τον ιδιοισμό της ότι αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά Λέει η Μαλάλα ότι η νέα γενεά αν δεν πάρει βιβλία και δεν εκπαιδευτεί θα πάρει όπλα και θα πολεμήσει. η κυρία Γκέριγκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στις 9 Οκτωβρίου ένα 14χρονο κορίτσι πυροβολήθηκε στο λαιμό και στο κεφάλι. Ήταν υπέρ της ε, εκπαίδευσης των κοριτσιών στα σχολεία. Οι Ταλιμπάν προανήγγυλαν ότι θα σκοτώνουν οποιονδήποτε παραβαίνει αυτές τις ε, διαταγές τους ε, και πηγαίνει στα σχολεία να εκπαιδευτεί. Βλέπουμε εδώ το τι συμβαίνει πέρυσι από ότι είχαμε ένοπλες ομάδες που εκατοντάδες επιθέσεις έκαναν εναντίον σχολείων. Πρόσφατα η πακιστανική κυβέρνηση ενέκρινε νομοθεσία ώστε να προστατεύονται τα σχολεία. Αλλά μέχρι να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία θα περάσουν χρόνια ολόκληρα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει το Πακιστάν και να ενθαρρύνει ώστε οι διεθνείς ε, προδιαγραφές ε, και κανόνες και κανονισμοί να τηρούνται. Όλοι οι πολίτες ε, θα πρέπει να έχουν τα ίδια ίσα δικαιώματα. Η κυρία Κίλν Νίσελεν έχει το λόγο. Εάν δεν δώσουμε μολύβια σε αυτή τη νέα ε, γενιά, τότε οι τρομοκράτες θα τους δώσουν όπλα. Αυτά ήταν τα λόγια της ε, Μαλάλα που καταπολεμά τον σκοταδισμό. Το 14χρονο αυτό κορίτσι αποτελεί προπομπό μιας κατάστασης τα νέα κορίτσια στο Αφγανιστάν ζουν αυτή την κατάσταση καθημερινά. Δεν ε, βεβαίως, δεν αποτελούν πρωτοσέλιδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορούν να απελευθερωθούν και να χειραφετηθούν οι Αφγανές γυναίκες. Δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Αυτό είναι το μήνυμα των βουλευτών από το Αφγανιστάν ε, λίγα, λίγες εβδομάδες ε, πριν φοβούνται ότι το 2014 όλα τα κεκτημένα θα ε, αρθούν και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτές τις δειλές πράξεις αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις τοπικές οργανώσεις γυναικών που θέλουν να κρατήσουν ανοιχτά τα σχολεία. Ευχαριστούμε την κυρία Κιλνίστελ από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές κυρία Νίκολ, ο κύριος Νίκολσον. Καταρχήν θα ήθελα αυτό το κορίτσι να ανανύψει σύντομα. Αυτό το κορίτσι έδειξε μεγάλο θάρρος στα 14 της χρόνια μίλησε για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει έμπνευση για όλους. Μιλάμε για 75 εκατομμύρια κορίτσια παγκοσμίως που στερούνται αυτό το δικαίωμα, το οποίο εμείς θεωρούμε δεδομένο. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα παιδιά στην εκπαίδευση. Αυτός είναι απότερος στόχος και είναι σαφές ότι σε πολλές χώρες αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα για τα κορίτσια. Στους στόχους της χιλιετίας θα πρέπει να δούμε και την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών όπως τη μαλάνα που απειλούνται σε καθημερινή βάση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απάνθρωπες συνέπειες. Ελπίζω χώρες όπως το Πακιστάν που δεσμεύτηκε ε, υπέρ των κοριτσιών και των γυναικών να το πράξει έμπρακτα να γίνει δηλαδή αυτό και όχι θεωρητικά. Ο κύριος Μπέλτερ έχει το λόγο για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ο συνάδελφος Νίκολσον, έτσι και εγώ ο ίδιος θα ήθελα να ευχηθώ καλή ανάρρωση, σιδερένια στην Μαλάλα Ιούσαυσάη. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να αναρρώσει μετά από τον σοβαρότατο τραυματισμό της. Και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ απογοητευτική αυτή η κατάσταση όταν βλέπουμε ποιο είναι το σύστημα ε, παιδείας και εκπαίδευσης. Η φτώχεια αναγκάζει αυτά τα παιδιά να καταλήγουν στα ιεροσπουδαστήρια, στους μετρεσέδες και καταλήγουν μετά στους Ταλιμπάν. Και αυτό είναι η ε, ακολουθεί μετά μια ε, στάση ακραία από πλευράς τους, ε, ιδιαίτερα εις βάρος των κοριτσιών. Γι' αυτό το σύνολο του συστήματος ε, παιδείας και εκπαίδευσης στο Πακιστάν δεν χρηματοδοτείται και επαρκώς ώστε να γίνει κάτι καλύτερο. Μόνο ένα σε κάθε τρία κορίτσια πάει στο σχολείο. αυτό πρέπει πραγματικά το θάρρος τους ε, να ε, τονωθεί ώστε και επιτέλους η κυβέρνηση του Πακιστάν να αναλάβει κάποια μέτρα, να κάνει κάτι. Και αυτό πρέπει να απευθυνθεί ως μήνυμα στο Ισλαμαμπάντ. Ευχαριστώ. Κυρία Ισάγια παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε δολοφονίες ε, από πλευράς των Ταλιμπάν και η περίπτωση προσπάθειας να δολοφονήσουν την ε, Μαλάλα Ιουσαφσάη μας συγκλονίζουν. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το θάρρος ε, αυτής, της, αυτού του κοριτσιού. Η κατάσταση των δικαιωμάτων των κοριτσιών είναι πραγματικά δεινή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να βελτιωθεί η κατάστασή τους και η κατάσταση των γυναικών στο Πακιστάν. Γίνεται προσπάθεια να έχουν δικαίωμα στην παιδεία και στην εκπαίδευση αυτά τα κορίτσια πολλές φορές δεν κατανοούν οι γονείς πόσο σημαντική υπόθεση είναι να πάνε στα σχολεία τα παιδιά τους και το ότι όταν πηγαίνουν τα κορίτσια στο σχολείο αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο. Μόνο 10-12% μπορούν να ε, ε, διαβάζουν ε, και έχουν μάθει τα σχετικά από τα μαθήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε το Πακιστάν να βελτιώσει την κατάσταση των παιδιών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καταδικάσω και εγώ την να καταδικάσω και εγώ την εξτρεμιστική πράξη κατά της Μαλάλα και πιστεύω ότι οι γυναίκες και τα νέα κορίτσια θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Θα πρέπει οι πακιστανικές αρχές να διασφαλίσουν αυτό το δικαίωμα. Δυστυχώς αυτή η βάρβαρη πράξη δείχνει ότι το καθεστώς ε, χρησιμοποιεί κάθε μέσο, το καθεστώς των ε, Ταλιμπάν και η Μαλάλα το μόνο που τόλμησε ήταν να αναφέρει στον ιστότοπό της, στην ιστοσελίδα της, την βία την οποία, στην οποία υπόκεινται τα νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη το Σύνταγμα το οποίο μιλά για το δικαίωμα στην εκπαίδευση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο δραστήρια για να καταδικάσει το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κρέτσου. Τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μακοβέη για ένα λεπτό. We as the European Union have an Θα πρέπει να προστατεύσουμε όλους τους πολίτες, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στα 27 κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε και τους πολίτες που δεν μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Μαλάλα ήταν ένα 14χρονο κορίτσι το οποίο ζήτησε το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτό ήταν το έγκλημά της. Και η κατάσταση καταδεικνύει την καταστολή όλων των δικαιωμάτων στο Πακιστάν. Περνάνε ε, νόμοι κατά της βίας προς τις γυναίκες και θα πρέπει να καταδείξουμε ότι αυτό δεν ε, επαρκεί. Το Πακιστάν είναι η τρίτη πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο για τις γυναίκες. Θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη δύναμη και να προωθήσουμε την ε, ανάπτυξη και τη βοήθεια έτσι ώστε να, υπάρχουν, να υπάρχει διασφάλιση δικαιωμάτων. Το Πακιστάν θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ασφάλεια των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου. Άσχετα με τη χώρα και τη θρησκεία θα πρέπει να εξασφαλίσει το δικαίωμα στην παιδεία για όλα τα παιδιά. Και οι διακρίσει ε, για λόγους φίλου θα πρέπει να καταδικάζονται και να στελιτεύονται. Οι δράσει των Ταλιμπάν στο Πακιστάν κλειδονίζουν την ασφάλεια στη χώρα και διακυβεύουν το μέλλον της. Μόνο το 2012 250 σχολεία καταστράφηκαν και 750 σχολεία υπέστησαν ε, σοβαρές υλικές ζημίες. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Θα πρέπει οι πακιστανικές αρχές να εξασφαλίσουν καλύτερη προστασία των σχολείων. Με απασχολεί ιδιαίτερα το πρόβλημα των επιθέσεων σε νέες γυναίκες που το μόνο που διεκδικούν είναι η μόρφωσή τους. Θέλουν να πάνε στο σχολείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θρησκεία που δικαιολογεί την απαγόρευση της πρόσβασης στην παιδεία των γυναικών. Οι πακιστανικές αρχές θα πρέπει να λάβουν κάθε μέτρο για να αποτρέψουν στο μέλλον τέτοιες ε, επιθέσεις και να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στην παιδεία των ανδρών και των γυναικών. Η κυρία Κάλεμπαχ παρακαλώ για ένα λεπτό με Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία ολόκληρη σειρά ε, λογοτεχνικών τοποθετήσεων για τη θέση των γυναικών στο Πακιστάν και κυρίως των κοριτσιών. Είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βλέπουν την κατάσταση εδώ και χρόνια, κυρίως στην Ήπεθρο ε, και έχουν περιγράψει πώς ακριβώς ε, εμποδίζονται τα κορίτσια να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση, πώς οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Και παρόλα αυτά θεωρείται αυτονόητο στο Πακιστάν οι γυναίκες να εξαρτώνται από τους άντρες συγγενείς τους. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση στο Πακιστάν όπου Υπάρχουν ε, γυναίκες που διεκδικούν δικαιώματα, όμως οι νόμοι που θεσπίζονται πρέπει να εφαρμόζονται. Στην περίπτωση της ε, Μαλάλα βλέπω να υπάρχει οργή και κραυγή κυρίως, κραυγή για να τους βοηθήσουμε. Εμείς λοιπόν καλούμεθα να εφαρμόσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν. Τα βήματα τα οποία γίνονται στο Πακιστάν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, αλλά κυρίως να παρακολουθούμε την εφαρμογή των νόμων. Ένα λεπτό κυρία Όγγιλαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε την διακήρυξη για την θρησκευτική ανεξαρτησία και την πρόσβαση των κοριτσιών στην παιδεία. Δυστυχώς, παρά τις διακηρύξεις αυτές, εξακολουθούν υπάρχουν εκφοβιστικές ε, και τρομοκρατικές ενέργειες ε, των Ταλιμπάν και αποτροπή των γυναικών από πρόσβαση στην παιδεία. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της Μαλάλα Σαπασάη και ε, να συστήσουμε στις πακιστανικές αρχές τα κόμματα να καταδικάσουν αυτή την επίθεση γιατί πραγματικά καταστρατεί κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες. Δεν θα πρέπει να επικρατήσουν οι ε, πολέμη το, της ισότητας των φύλων και οι τρομοκράτες. Ο κύριος Στάνοκ. Σίγουρα ήταν αποτρόπαιο το έγκλημα της, κατά της Μαλάλα. Ένα 14χρονο κορίτσι που το μόνο της α, ε, λάθος ήταν ότι διεκδίκησε πρόσβαση στην παιδεία. Κρίμα που οι πακιστανικές αρχές δεν μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες από τέτοιες αποτρόπες ενέργειας. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες, τέτοια ιστορικά ε, κατά ε, ακόμη και υπουργών που ε, απειλήθηκαν επειδή προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τέτοια ισότητα. Δύσκολο μπορούμε να βρούμε λόγια για να καταδικάσουμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Βέβαια, είχαμε κατακραβεί παγκόσμια ε, και τις φωνές στο Πακιστάν που υψώθηκαν ε, εκφράζοντας ε, την οργή και την αντίσταση στο πεπρωμένο της Μαλάλα. Χαίρομαι γιατί είμαι υπερήφανος που υπάρχει κάποια προσπάθεια ευελτίωσης και ανάνυψης ε, της Μαλάλα χάρη στις προσπάθειες της υπεράνθρωπης προσπάθειας των γιατρών στο Μπέρμιχαμ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ επιθυμώ να εκφράσω την υποστήριξή μου προς αυτή την έφηβο η οποία έγινε το σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων γυναικών. Η Μαλάμα είναι μόνο 14 ετών, είναι όμως πολύ θαραλέα και γι' αυτό λοιπόν έγινε φόβος και τρόμος των Ταλιμπάν τα δικαιώματα των γυναικών, ε, το δικαίωμά τους ε, στην εκπαίδευση αποτελεί και τρόμο για τις Ισλαμικές ε, κοινωνίες γενικότερα. Αυτό βέβαια δεν μας εκπλήσει. Εκείνο που μας εκπλήσει είναι ότι οι κοινωνίες αυτές είναι τόσο προχωρημένες έχουν φτάσει στο σημείο να δίνουν όπλα σε παιδιά ηλικία 14 ε, ετών και μικρότερα. Αυτά τα παιδιά βέβαια χρειάζονται εκπαίδευση και τούτο ε, αποδεικνύει ότι οι Ταλιμπάν αποδυναμώνται τη στιγμή που θέλουν ε, να καταπιέσουν τέτοιου είδους δικαιώματα. Επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω Τέτοιου είδου περιπτώσεις ε, μας κάνουν να σκεπτόμαστε κατά πόσον η πολυμορφία και η πολυεθνικότητα είναι η σωστή πολιτική όχι. Νομίζω ότι απέτυχε ο πολυπολιτισμός. Στην περίπτωση αυτή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δέχτηκε οξύτατη επίθεση. Και εκεί νομίζω ότι σταματάει η συζήτηση περί ισότητας. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να καταπολεμούνται. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει επίτροπος Γκέγαν Κουίν. Ευχαριστώ. Κύριε, η είπατε εκπρόσωπος ε, ε, Άστον φυσικά καταδικάζει και στυλιτεύει την τον πυροβολισμό και την επίθεση κατά της Μαλάλα στις 9 Οκτωβρίου από εξτρεμιστές. Θεωρεί ότι είναι αποτρόπη η επίθεση και κατάφορη παραβίαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και πλήγμα κατά των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν. Πάντως ε, είναι αισιόδοξη η κατάσταση της υγείας της ε, Μαλάλα στο Μπέρμιχαμ και όλοι της ευχόμαστε καλή ανάρρωση και σύντομη ανάνυψη. Οι Θελιμπάν του Πακιστάν αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να τη σκοτώσουν αν αναρρώσει. Θα πρέπει οι πακιστανικές αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της Μαλάλα και της οικογένειάς και άλλων που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες απειλές. Η Μαλάλα διεκδίκησε εφαρμογή των δικαιωμάτων παιδείας και για τα κορίτσια και ήταν πολύ θαραλέα η δράση της. Ε, μπορούμε, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε για το κουράγιο της αυτή, τη, αυτή την κοπέλα. Σίγουρα έχουμε την παιδεία ως προτεραιότητα στη σχέση μας με το Πακιστάν. Ιδιαίτερα το θέμα της επαγγελματική κατάρτισης μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στην παιδεία και την κατάρτιση και για τα κορίτσια. Θέλουμε να συνεργαστούμε με το Πακιστάν για να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα στηρίζεται στην ενοχή. Τα θέματα ισότητας ε, των γυναικών και των παιδιών ε, πολύ τακτικά ε, επισημένονται στον Διάλογο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκή Ένωση Πακιστάν. Και μάλιστα στην πρόσφατη αποστολή που είχαμε είπατε εκπρόσωπο πως ε, στο Ισλαμαμπάτ στις 6 ε, Ιουνίου επισήμανε και πάλι το θέμα αυτό. Ενθαρρύναμε την κυβέρνηση του Πακιστάν να αναλάβει κατεπηγόντως μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Επιπλέον, Προβλέπουμε ε, χρηματοδότηση για ανθρωπιστικά προγράμματα, για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας, την πάταξη της διακριτικής μεταχείρισης βάρος, βάρος παιδιών και γυναικών, πρόσβαση στη δικαιοσύνη και άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Σημαντικά νομοσχέδια έχουν ε, εγκριθεί και θα συνεργαστούμε στενά με τις επαρχίες που τώρα πια έχουν εκτεταμένες αρμοδιότητες για όλα αυτά τα θέματα. Πάντως μας ανησυχεί σοβαρά ε, η βλάβη που φέρνει αυτό το κλίμα εκβοβισμού ε, στην ανάπτυξη του Πακιστάν. Θέλουμε να ενισχύσουμε το διάλογο που υπάρχει με τακτικούς τομέακους διαλόγους για την ασφάλεια, για το κράτος δικαίου, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αντιμετώπιση τη εξτρεμιστική βία ε, θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα του διαλόγου αυτού. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μα με το Πακιστάν στο μέλλον. Η υποστήριξη των δημοκρατικών θεσμών του Πακιστάν και της κοινωνίας των πολιτών του Πακιστάν θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο αυτής της συνεργασίας. Το περιστατικό της 9ης Νοεμβρίου οδήγησε κατακραυγή στην πακιστανική κοινωνία. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά είπε ότι το Πακιστάν δεν θα πρέπει να επιτρέψει ε, να τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών τους ε, από μια τέτοια κατάσταση και θα πρέπει να απαταχθεί ο εξτρεμισμός. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους ηθήνοντες του Πακιστάν που θέλουν να πατάξουν την τρομοκρατία και την ιδεολογικά υποκινούμενη βία να επικρατήσουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ. Έχουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος. Θα ψηφίσουμε στις 11.30. Και περάμε στην κατάσταση Καμπότζη. Για ένα λεπτό το λόγο κυρία Γκόμες